2 ε, τα μέλη ή πολιτικές ομάδες ε, που είναι, που είναι τουλάχιστον τον ε, μέσο, στο μέσο όριο θα μπορούν μέχρι αύριο 27 Απριλίου στις, τα μεσάνυχτα να υποβάλουν την απόφασή τους να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Εάν δεν υπάρξει αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για αυτή την απόφαση θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις τους ε, απευθείας. Θα ήθελα να σας ενοκοινώσω ότι σύμφωνα με το τον ε, άρθρο 46.2 του κανονισμού ε, δέχτηκα δύο προτάσεις για ε, νομοσχέδιο ε, της Ένωσης. Μία πρόταση για τις διαφορετικές δηλώσεις, τη σύσταση και τη γεύση των προϊόντων στην κεντρική και ανατολική και δυτική αγορά της Ένωσης που υπέβαλε η κυρία Σουίτσα και εννέα άλλοι μέλη. Πρόταση έπειτα για έναν άλλο κανονισμό όσον αφορά τον έλεγχο για τις εξωτερικές ε, τις αλλοδαπές επενδύσεις τραγικού τομεί που έχει υποβάλει ο κύριος Δανιέλ Κάσπαρη και οι προτάσεις αυτές παραπέφθηκαν σε αρμόδιες επιτροπές.